για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Ορισμένοι εξ αυτών βρίσκονται σε μια κατάσταση επικίνδυνη και οφείλουμε να θυμίσουμε ότι η βουλευτής Λέιλα Ζάνα που κέρδισε το βραβείο Ζαχάροφ το 1995 μόλις ε, αφαιρέθηκε από βουλευτή τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση στο Ευρωκοινοβούλιο, θα ήθελα να τη εκφράσει την αλληλεγγύη όλων των Ευρωβουλευτών, γιατί δεν είναι αποδεκτό σε μια δημοκρατία ένα ε, κλεγμένο εκπρόσωπο του λαού να καθερείται ε, παράνομα. Θέλω δε να εκφράσω. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Θέλω δεν να εκφράσω την ανησυχία μου για τις επανειλημμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία εις βάρος όχι μόνο των αντιφρονούντων αλλά και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι και ε, ε πανεπιστημιακοί. Να θυμίσω τον Ρέι Γκούλμεν, Σεμίο Τζάσκα, Οσμάν Καβαλά, Μεμέτα Τάν και Σαΐν Αλτάι το Ευρωκοινοβούλιο δεν θα παραλείψει να εκφράσει την στήριξή του στους αγώνες αυτών των ανθρώπων υπέρ της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. οπω γνωρίζετε, το πρωί μετά από την παρουσίαση